Ε, Συνάδελφοι, έλαβα από το Συμβούλιο τις θέσεις που υθετήθηκαν στην πρώτη ανάγνωση και τους λόγους οδήγησα στο Συμβούλιο να θετήσει αυτή την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά δημοσιευτούν στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Ε, έχει, έχει τρεις μήνες το Κοινοβούλιο ε, που ξεκινά από αύριο το Κοινοβούλιο. Από αύριο 3 Απριλίου του 2014 ξεκινάει περίοδος ε, της οποίας θα πρέπει να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση Ζαλεύσκη όσον αφορά την μείωση ή την κατάργηση των τελωνιακών δασμών στα εμπορεύματα που προέρχονται